Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου. Επί της έκθεσης ε, Βόρτμαν Κόλ. Το λόγο έχει η κυρία Μανέσκου για ένα λεπτό. υπέρ. Ψήφισα υπέρ του Six γιατί έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να παγιώσουμε την χρηματοπιστωτική πειθαρχία για να πετύχουμε τους στόχους μας αυξημένη ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουμε τις, ε, τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να αναλάβουμε έντονες ε, δεσμεύσεις η εμπειρία που έχουμε τα δέκα τελευταία χρόνια τονίζουν την ανάγκη για οικονομική και ε, χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε πιο δεσμευμένοι και να έχουμε καλύτερες μεθόδους επιτήρησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό χρειάζονται απαραίτητα πρότυπα για τους προπολογισμού και ταυτόχρονα να έχουμε αποτελεσματικές ε, χρηματοπιστωτικές διαδικασίες. Οι προπορισμοί θα πρέπει να βασίζονται σε σωστές ε, διαδικασίες. Ο κύριος Μαστέλα έχει το λόγο. Ε, Απόν. Ο κύριος Μπαλντασάρ έχει το λόγο, ένα λεπτό. Ποιος Τρεις, Απόν. Ο κύριος Σούστα, λοιπόν, έχει το λόγο. Grazie, Presidente ψήφισα υπέρ της έκθεσης Βόρτμαν Call και νομίζω ότι σε ε, μια τέτοια δύσκολη χρονική στιγμή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε με σπουδή στο αίτημα των πολιτών. Αυτό το παρκέτο το κρίνω ανεπαρκές. Όμως είναι απόλυτα αναγκαίο να συνεχίσουμε ακολουθώντας αυτή την οδό της ανάπτυξης και των δημοσιονομικών ελέγχων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα την αναπτυξιακή πορεία. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η Ένωση. Αυτή είναι μια πρώτη απάντηση και δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία γιατί εδώ και χρόνια δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε με την κατάλληλη ταχύτητα στις ε, κρίσεις. Η κυρία Ματέρα για ένα λεπτό. Απούσα η κυρία Ματέρα. Το λόγο έχει ο κύριος Γιάρ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο τίτλος μιας μια εφημερίδα στη Γερμανία ήταν ότι ο Τίγρης αποκτά δόντια. Ενδυναμώνεται η θέση τη Κομισιόν. Μπορούσα λοιπόν να υπερψηφίσω γιατί ακριβώς αυτό έγινε όσον αφορά και τον περιορισμό των ελλημάτων όσον αφορά τα προβλήματα, ότι θα υπάρχει ημιαυτόματος μηχανισμός κυρώσεων ούτως ώστε μετά το 2012 να ελέγχουμε τις ανισορροπίες και μακροοικονομικά. Αυτά είναι σημαντικά βήματα σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Κομισιόν έκανε ό,τι πρέπει για να μπορέσει να σταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ζώνη ευρώ. Αυτό που μας λείπει είναι η ενεργή συμμετοχή των κρατών μελών και θέλω να παρακαλώσω τα κράτη-μέλη να ε, συμπλέψουν με αυτές τις συντονιμένες δράσεις και να πάρουν αποφάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιάρ. Το λόγο έχει ο κύριος Ούτζα, η κυρία Ματέρα. Η οποία καθυστέρησε θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε μεγάλες δυσχέρειες στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό χρειάζεται μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση μια κοινοτική εποπτεία που να είναι πιο σταθερή και συνεχής σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές. Αυτό αφορά την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και παραγωγικότητα καθώς και απασχόληση. Γι' αυτό θα πρέπει να εγκριθεί αυτό το πακέτο έξι νομοθετημάτων έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε μία επαρκή δέσμευση για τη σταθερότητα των οικονομιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Για ένα λεπτό ο κύριος Ούτζας έχει το λόγο. Ψήφισα υπέρ του πακέτου των έξι νομοθετημάτων γιατί έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να ελέγξουμε τους προϋπολογισμούς και τα δημοσιονομικά μας εκεί όπου απέτυχαν τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό το θέμα αφορά την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η Ευρώπη αναλαμβάνει συγκεκρινήσεις έναντι των πολιτών για μια σταθερότητα, για μια οικονομική διακυβέρνηση και για μια ανάπτυξη, ένα ρυθμό ανάπτυξης, γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχει μέλλον για τους πολίτες και για τις μέλουσες γενιές. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ. Και εγώ υποστηρίζω αυτό το ε, νομοθέτημα του πακέτου των ε, έξι νομοθετημάτων, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και ενωμένοι και για θέματα οικονομικής διακυβέρνησης και για θέματα συνοχής, ενδοκινοτικής συνοχής. Θα πρέπει να ελέγχουμε τα κράτη-μέλη και το συντονισμό τους και περιμένουμε από όλα τα κράτη-μέλη να προβάλλουν συγκεκριμένα μέτρα μέσα στα πλαίσια ενός έκτακτου σχεδίου για τον ανταγωνισμό και την πραγματική απασχόληση για, για τον ε, μη κοινωνικό αποκλεισμό των φτωχών. Αυτό, σε αυτό στοχεύουμε για τους επόμενους έξι μήνες. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Απούσα. Ο κύριος Καρόνα για ένα λεπτό. Ζούμε μία ε, δυσχερή κατάσταση ως προς το μέλλον του ευρώ. Έχοντας ε, πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος, θα έπρεπε να περάσουμε σε μία πολιτική πλήρους ελέγχου των δημοσιονομικών των κρατών μελών, γιατί θέλουμε να μειώσουμε και το έλλειμμα και το χρέος. Χωρίς μια ευφύ πολιτική επενδύσεων που θα μπορέσει να δώσει μια νέα πνοή στις οικονομίες, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι πλέον φτωχοί θα καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Γι' αυτό καταψηφίσαμε οι περισσότεροι σοσιαλιστές αυτή την έκθεση, διότι η λιτότητα χωρίς ανάπτυξη είναι μία εντελώς λανθασμένη πορεία και οδός. Η κυρία Χάρκιν, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χθες πολλοί από εμά είδαμε μια ε, μια βιντεοτενία πώς μπορεί κανένας να κερδίσει από μια πτώχευση πως ε, οι άλλοι άνθρωποι χάνουν ε, τα χρήματά τους αυτός ο, ο προδότης αν θέλετε που είχε κάνει αυτό το, τη βιντεοτενία μας είπε ότι δεν έφταναν οι κυβερνήσεις έφταιγε η Goldman Sachs και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τη σωστή προσέγγιση. Εγώ αρνούμε εγώ και οι Ιρλανδοί ε, εκλογή να δώσω ισχύ στις αγορές. Δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Είμαστε μέλος ενός κακά οργανωμένου ε, νομίσματος, αλλά θα πρέπει τα παλιά ε, σφάλματα να έχουν επίδραση στις εξελίξεις του μέλλοντος. Ε, λέμε βέβαια ότι βάζουμε το, κλείνουμε το πηγάδι μετά που έχει πέσει το μωρό μέσα, αλλά αυτή η έκθεση κατά μένα είναι μονάχα ένα λίγο οξυγόνο, δεν είναι η θεραπεία του προβλήματος. Ευχαριστώ κύριε Χάκη. Ένα λεπτό, ο κύριος Καρίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Ευρώπη έχουμε μια χρηματοπιστωτική θύελα, κρίση εμπιστοσύνης. Οι αγορές δεν εμπιστεύονται τα κράτη-μέλη γιατί δεν πιστεύουν ότι τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρήματα που έχουν ήδη δανειστεί. Σήμερα το Six Pack για την χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική εποπτεία που επεξεργαστήκαμε και εγκρίναμε είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα πρόοδου ώστε να σταματήσει η θύελα, να ανακτήσουμε την αξιοπιστία των αγορών προς τις εθνικές κυβερνήσεις και οικονομίες και για την ευμερία των λαών μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όμως, ας θυμηθούμε ότι αυτά θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα, αλλά η Κομισιόν εξακολουθεί να πρέπει να κάνει πολλά πράγματα τώρα πρέπει να μας δώσει ένα σχέδιο πιο σαφές για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σουάμπ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος ότι το κλειδί της στρατηγικής ε, θα πρέπει να βρεθεί τώρα για μια στρατηγική δηλαδή που τελικά θα ενδυναμώσει τελικά την Ευρώπη να βγει πιο ισχυρή από την κρίση από την πήγε στην κρίση. Το σημαντικό θέμα θα ήταν κατά πόσον τα μέσα που αποφασίζονται μέσα στα πλαίσια του Six Pack, ιδίως στις εκθέσεις Βόρτμαν ε, Κόλ και Φάγιο, επιτρέπουν αυτού του τύπου τον έλεγχο. Ο συμβασμό που επιτέχθη τώρα όσον αφορά το προληπτικό τμήμα του Συμφώνου Σταθερότητα ε, προβλέπει δύο βήματα. Καταρχήν, το Συμβούλιο μπορεί κατόπιν ε, προτάσεις Κομισιόν να ψηφίσει με σταθμένη πλειοψηφία για την διόρθωση της μακροοικονομίας ενός κράτους μέλους. Η πρόταση αυτή μπορεί να ξαναποβληθεί από την Κομισιόν σε ένα μήνα αν δεν έχει δράσει το Συμβούλιο και μπορεί να απορριφθεί τη δεύτερη φορά αυτόματα εάν δεν, μάλλον να εφαρμοστεί αν δεν έχει απορριφθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο τα κρατη θα τηρήσουν αυτά που ε, θα τους επιβληθούν ή θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τους κανόνες όπως το 2003. Εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να επικρατήσει η κοινοτική μέθοδος και να μπορούσαν τελικά αποτελεσματικά να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σουάπ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις αγορές. Αυτή είναι η μακροχρόνια απάντηση στην κρίση. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπονται μακροπροληπτικά μέτρα και με μία πλειοψηφική ψήφο και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ε, διεθνική και εθνική διαχείριση παράλληλα. Εγώ ψήφισα υπέρ της ολοκλήρωσης αυτής για να υπάρξει σύγκληση και μία πραγματική οικονομική και νομισματική πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές κρίσεις Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Πολωνική Προεδρία καθώς και την Ουγγρική. Ευχαριστούμε κύριε Μεσάρος. Ο κύριος Χάναν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Μετά την κρίση, τι γίνεται, έχουμε μεγαλύτερο χρέος και μεγαλύτερο έλλειμμα. Δεν υπάρχουν πλέον κρατικά κονδύλια. Και τώρα Εφόσον δεν μπορούμε να προστρέξουμε ούτε στην ΕΚΤ, τι κάνουμε. Ζητάμε ε, την, ε, ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι τραπεζίτες ζητάνε να περάσει το κόστο να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Πού γίνονται περισσότερες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στο City, όμως ε, αποστέλλεται ο λογαριασμός για ένα κοινό νόμισμα για ένα κοινό νόμισμα στο οποίο εμείς δεν θέλουμε να προσχωρήσουμε. Το ίδιο γίνεται και με την ΚΑΠ, καθώς και με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Και τι γίνεται. Πρόκειται για ε, ένα κυκλόπιο τείχος το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, διότι δεν μπορούν οι πολίτες να καταβάλουν εσαΐ το κόστος και πιστεύω ότι θα διανύσουμε και μία νέα κρίση. Θα διανύουμε αλλεπάλληλες κρίσεις που θα πρέπει να... Ε, όπου και πώς έλεγε ο, ο Σέξπιρ, οι κρίσεις διαδέχονται μια φορά σήμερα. Χάρηκα πολύ που υποστήριξα το Six ΠΑΚ. Στη δημοκρατία οι κυβερνήσεις και η αντιπολίτευση ε, εξαγοράζουν εκλογές αν τους μπορούν να τα καταφέρουν και βεβαίως η στάση είναι μην πληρώνει σήμερα αυτό που μπορείς να αναβάλεις για αύριο. Αυτή η υπερβολή εν μέρη τουλάχιστον μας οδήγησε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευτυχώ έχουμε αρχίσει κάτι να κάνουμε και να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και όπως είπε ο συνάδελφος Μάρτιν Χάρτ η πολιτική υποτίθεται ότι είναι αυτοί που ελέγχουν τα πράγματα και όχι οι αγορές η οικία αξιολόγηση. Οπωσδήποτε αυτό σημαίνει ότι κάναμε έξι βήματα πρόοδου. Ο κύριος Κέλλη τελείωσε. Ο κύριο Σιλβέστρης, ευχαριστώ και εμείς ψηφίσαμε υπέρ του πακέτου έξι νομοθετημάτων. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με μία πορεία για την καλύτερη κοινή οικονομική διακυβέρνηση. Πρόκειται για ένα βήμα αποφασιστική αποφασιστικής σημασίας και δεν μπορούμε να μην γνωρίζουμε τι έχασε η Ευρώπη. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στις 16 Ιουνίου ο πρόεδρος Πανοροπόη μας μίλησε εδώ για την ανάγκη του να μιλάμε για την, όχι για την Ευρωζώνη, αλλά για την Ευρωχώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μπαρόζο ήταν ιδιαίτερα οξυδερκή σήμερα και, αλλά το 2008 μας είχε πει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την ύφεση. Μιλάμε για μία ευρωπαϊστική συμφίση-νένεση, αλλά πρόκειται στην ουσία για μία οικονομική διακυβέρνηση και μία πολιτική που αναλαμβάνει ε, ευθύνες για την ανάπτυξη χωρίς να επιτρέψει την κερδοσκοπία των αγορών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιλβέστρης. Περνάμε στην έκθεση Γκουλάρ. Και το λόγο έχει ο κύριος Μπαλτασάρε. Mm. Πρόεδρε, η κρίση δείχνει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έξι κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα ισολογισμού και μπορούν να βρεθούν σε κατάσταση ε, μη ανταπόκριση στο χρέος και πάυσης πληρωμών. Γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση Γκουλάρ, όπου θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται δόλιος χειρισμός στατιστικών στοιχείων από κράτη-μέλη. Παράλληλα όμως θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες αποτροπής προβλημάτων, δηλαδή μια πραγματική ονέ. Οι κυρώσεις θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τα κράτη, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν νομίμως και θα υπάρχει μια πραγματική εποπτεία και με τη βοήθεια των ευρωομολόγων. Ευχαριστούμε κύριε Καλτασάρε. Η κυρία Αντζελίλη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την έγκριση του πακέτου έξι νομοθετημάτων το Κοινοβούλιο ανοίγει το δρόμο για μια πραγματική στρατηγική έναντι της ε, κρίσης. Μιλάμε για διαφάνεια προϋπολογισμών, μείωση του χρέους, αλλά όπως είπε χτες και ο Γιούνκερ και επανέλαβε σήμερα ο Παρόζο, θα πρέπει να σταθούμε στην ανάπτυξη. Έχουμε mm. να διανύσουμε μακρύ δρόμο και σήμερα ο Μπαρόζο μας μίλησε για τα μελλοντικά βήματα μιας ε, θαρετής στρατηγικής Μιλάμε για μια σειρά προτάσεων για τα ευρωμόλογα και για έναν φόρο στις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Μιλάμε για 56 δις ευρώ έσοδα μόνο από αυτό το φόρο γιατί θα πρέπει οι τράπεζες ε, να, και οι τράπεζες να υποστούν το κόστος της ε, κρίσης και όχι μόνο οι πολίτες. Ο κύριος και έχει το λόγο. Ο κύριος θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω διότι αυτός ο κανονισμός δεν είναι μόνο σημαντικός για την Ευρωζώνη. Πρέπει να πω ότι είναι σπουδαίος και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το βασικό πρόβλημα είναι το συνεχιζόμενο έντονο ενδιαφέρον ε, ώστε να πιεστούν τα κράτη τα οποία δεν προχωρούν στην εξυγίανση των ε, προϋπολογισμών. Δηλαδή η ανοχή οπωσδήποτε τελικά οδηγεί σε μεγάλες κρίσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει κανείς από αυτές τις χρήσεις και το τίμημα είναι και πολύ ψηλό. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε λοιπόν ε, διατάξεις οι οποίες είναι μια καλή απαρχή. Τονίζω όμως ότι αυτό είναι το μόνο, μόνο το πρώτο βήμα. Χρειάζεται περισσότερη πειθό και επιμονή για να εκτελεστούν σωστά οι πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο, κύριος... ο κύριος Σούτζας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο Σιλβί Κουλάρ γιατί έφερε σε αίσιο πέρας αυτό το σημαντικό ζήτημα και θέμα. Μιλάμε για μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πρόκειται για μια πράξη που οδηγεί, που φέρει σε πέρας τις δηλώσεις που ακούσαμε και σήμερα στην αίθουσα αυτή, που όμως δεν τίθενται σε εφαρμογή έμπρακτα. Όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις αρχής όλοι συμφωνούμε. Όταν ψηφίσαμε το πρόγραμμα της Επιτροπής θα έπρεπε να, τεθεί σε εφαρμο... σε εφαρμογή. Και αυτό που έχει σημασία είναι να τεθεί σε εφαρμογή έμπρακτα αυτό το πρόγραμμα. Το λόγο έχει η κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα την έκθεση της Σιλβί Γκουλάρ όπως και άλλες ε, εκθέσεις που αναφορούν στο six pack δεν είναι ο σκοπός να λυθεί το τρέχον πρόβλημα. Ένα μέρος αυτού του προβλήματος παρουσιάστηκε σήμερα από τον κύριο Μπαρόζο, αλλά νομίζω ότι έτσι για πρώτη φορά έχουμε κάποιες ελπίδες. Ε, που έχουν σωματωθεί στην σύγχρονη πραγματικότητα. Όσον αφορά όμω αυτή την έκθεση, με χαρά μου είδα ότι περιελήφθηκε το άρθρο 9 που λέει ότι η Ένωση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις υποχρεώσει τη που σχετίζονται με την υψηλή ανεργία, την επαρκή κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ωραία λόγια βέβαια, αλλά εμεί έχουμε την ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταφραστούν σε πραγματικότητα. Επίση χαίρομαι που υπάρχει ευελιξία σε αυτή την έκθεση όπου αναφέρεται ότι το Συμβούλιο ε, θα μπορούσε να αποφασίσει να μειώσει τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε ένα κράτος μέλος μετά από αίτηση, ε, ε πρόταση της Κομισιόν και μετά από δικαιολογημένη αίτηση του κράτους μέλους. Αυτό το είδους η ευελιξία είναι πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη και σε αυτό το πλαίσιο και για τη δική μου χώρα την Ιρλανδία. Ευχαριστούμε κυρία Χάκεν. Ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη συζήτηση που έγινε σήμερα το πρωί ο κύριος Μπαρόζο ανέφερε ότι θα ανεβεί μέχρι το 2020 ο αριθμός των ε, ε, απασχολούμενων ε, που απασχολούνται από το 67% στο 75%. Μα γιατί όχι 90% ε, οι ανακοινώσει των πολιτικών ε, σκοτίζουν οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα. Ε, πριν από το καλοκαίρι η κρίση είχε κηρυχθεί τελειωμένη. Οι αγορέ δεν πήραν όμω το μήνυμα και ο κύριο Μπαρόζο έγραψε στον Guardian ένα άρθρο που έλεγε ότι παρεξενευόταν. Ήταν έκπληκτο από την ε, συμπεριφορά των αγορών. Πώ ε, ε, οι αγορέ στην Ισπανία ή στην Ιταλία δεν άκουσαν αυτά που έλεγε η Κομισιόν. Αυτή είναι η ιστορία. Οι άνθρωποι κάνουν τα λάθη του. Αλλά εμείς ε, δεν θα πρέπει να ε, τραβηχτούμε μέσα στο ενιαίο νόμισμα. Το πρόβλημα με το six pack είναι ότι δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Εμείς είμαστε, ε, όπως είπε ο Τζόρτζιλ, ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε αλλά όχι να απορροφηθούμε. Θα πρέπει να απαντήσουμε όχι. Σας ευχαριστώ κύριε Χάναν. Η κυρία Κάινεν, παρακαλώ για ένα λεπτό. Arvoisa eh, eh, eh, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι με ικανοποίηση άκουσα τον λόγο του κυρίου Μπαρόζο. Έδειξε ηγετικό πνεύμα και υιοθετούνται τα αναγκαία μέτρα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και αυτά που χρειαζόμαστε για την Ευρώπη στο μέλλον. Χαιρόμαστε που και το Κοινοβούλιο υιοθέτησε από πλευρά του και τα μέτρα των προτάσεων six pack. Χάρη σε αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή βήματα προς μια κατεύθυνση ώστε να υπάρχει η σωστή ευθύνη και λογοδοσία και διαφάνεια από πλευρά της κοινότητας όπως απαιτείται και χρειάζεται σε σχέση με τα οικονομικά όπως ακούσαμε από τον κύριο Μπαρόζο και επίση ε, και από προηγούμενε τοποθετήσει, αυτά τα μέτρα αυτών δεν επαρκούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν μελλοντικά πακέτα δέσμες ε, για τις χρηματοοικονομικές αγορές και πρέπει περαιτέρω μέτρα να ληφθούν για να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Σας ευχαριστούμε. Και σε σχέση με την έκθεση Χαγκλόντ για ένα λεπτό θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ντεάντζελης παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εμπειρία αυτών των ετών μας λέει ότι είναι απαραίτητο ένα ενισχυμένο πλαίσιο ε, οικονομική διακυβέρνηση όπω είναι απαραίτητο να διευρυθεί και να ενισχυθεί το πλαίσιο τη εποπτείας και να γίνει αποτελεσματικό και αξιόπιστο με κυρώσει που θα μπορούσαν να αποτελούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό χαρακτήρα, ιδίω αν είναι ε, πραγματική η εφαρμογή του. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση ε, όχι μόνο μέσω ε, σχεδίων ε, λιτότητας. Αυτό δεν αρκεί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Και για το λόγο αυτό, για την έκθεση ε, Χαγκλούντ, απέσχον. σα ευχαριστούμε κύριε Ντάντζελε. Θα λάβει τον λόγο τώρα ο κύριο Αντωνιώτση, παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με την έκθεση αυτή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πόσες καινούριε και σημαντικές εξουσίες δίνει η συνθήκη της Λισαβόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτάσεις της Κομισιόν για μια καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση έχουν αποφασιστική σημασία για την οικονομική μας ανάπτυξη και ιδιαίτερα ε, για την ε, Ευρωζώνη. Οι βελτιώσεις για τη δημιουργία ενός ε, στέρεου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης είναι προφανής. Ε, συμφωνώ με τις γενικές θέσεις αυτής της έκθεσης και γι' αυτό ψήφισα υπέρ. Έχουμε νέες ευθύνες μπροστά μας. Το πακέτο των μέτρων θα βελτιώσει ε, περαιτέρω και θα ενισχύσει τις ευθύνες μας αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία ε, στις μακροοικονομικές, ε, ε, δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές και στον ιδιαίτερο ρόλο που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της εποπτείας και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν συχνές τακτικές δημόσιες ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνιώτση. Ο κύριος Ουτζίας τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαίρω κι εγώ τον συνάδελφο Χάγκλουντ για την εργασία που πραγματοποίησε και την οποία υπερψήφισα. Όπως και ολόκληρο το πακέτο. Ψήφισα υπέρ. Η έκθεση αυτή προβλέπει κυρώσεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι κυρώσεις που θα ε, επιβληθούν μόνο αν ένα κράτο μέλος αποδεικνύεται ότι δεν είναι διατεθειμένο να ε, εφαρμόσει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Γιατί αν δεν βελτιωθούν οι δημοσιονομικέ συνθήκες, κύριε Ντεάντζελης, δεν υπάρχουν δυνατότητε ανάπτυξη. Ε, όποιες και αν είναι οι προσπάθειες για ανάπτυξη δεν θα οδηγήσουν πουθενά, θα ακυρωθούν αν δεν υπάρχει δημοσιονομική εξυγίανση. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το πακέτο που θα ψηφίσουμε σήμερα θα είναι η βάση για να έχουμε αυτή την ανάπτυξη στην οποία θα πρέπει να στοχεύσουν όλα τα κράτη. Αν σταματούσαμε εδώ, δεν θα είχαμε επιτύχει φυσικά τους στόχους που θέτουμε, αλλά με το βήμα αυτό μπορούμε σίγουρα να επιτύχουμε και αυτόν αυτό τον άλλο στόχο. Ευχαριστούμε κύριε Ουτζίας. Ο κύριος Μέρφυ παρακαλώ. ευχαριστώ. Αυτά που ψηφίσαμε αποτελούν τη θεσμοποίηση της μόνιμης λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το πρόγραμμα επιτήρησης η Κομισιόν έχει οριστεί τώρα σαν χωροφύλακας ολόκληρης της Ευρώπης και τη στιγμή μάλιστα που χώρες που τολμούν να παραβιάσουν τη δημοσιονομική ορθοδοξία θεωρούνται σαν χώρες απίστων ή αμαρτωλές. Έτσι η εργατική τάξη πληρώνει για την οικονομική κρίση για την οποία δεν ευθύνεται η ίδια. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά για να δούμε ότι αυτά τα μέτρα λιτότητας είναι αποτυχημένα εκ των προτέρων. Δέστε τι γίνεται στην Ελλάδα, πόσο συρρυκνώθηκε η οικονομία. Δέστε την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Τα μέτρα λιτότητας έχουν ήδη αποτύχει και θα αποτύχουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέρφη. Τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Χάρκιν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστήριξα την έκθεση του Καρλ Χάγκλουντ που μας λέει ότι η πείρα που έχουμε ε, συγκεντρώσει τα τελευταία δέκα χρόνια δείχνει την ανάγκη που υπάρχει για, για οικονομική διακυβέρνηση με κοινού ε, κανόνες και ισχυρότερη εποπτεία. Αλλά δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Είτε πρόκειται για ευρωομόλογα ή ομόλογα σταθερότητας ή οτιδήποτε άλλο, ε, χρειάζονται και άλλοι μηχανισμοί για την υποστήριξη της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το πακέτο που ψηφίσαμε σήμερα θα λύσει τα προβλήματά μας, αλλά είναι μέρος μιας συνολικότερης ε, λύσης. Έχω ανάμεικτα αισθήματα αυτή τη στιγμή. Ένα μέρος αυτής της έκθεσης ε, έχει πραγματικά περιλαμβάνει σοβαρά μέτρα. Αλλά από την άλλη μεριά οι πολίτες περιμένουν να λειτουργήσουν τα συστήματα και προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί δεν θα είναι αυτό το πακέτο η λύση, αλλά θα συμβάλλει. Σε ευχαριστούμε Μπάτεν παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το λεγόμενο six pack ε, επιβάλλει επιτήρηση στα κράτη-μέλη από την Κομισιόν. Την εποχή του βασιλέως Εδουάρδου του πρώτου στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας είχε δηλωθεί ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας τα δημοσιονομικά και το 1642 ε, καθορίστηκε ότι μόνο το κράτος έχει το δικαίωμα να παίρνει φόρους, να εισπράττει φόρους. Αυτή τη στιγμή όμως η Βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να δεχτεί τέτοιο δημοσιονομικό έλεγχο από έξω από την Κομισιόν. Αν το πράξει τότε δεν μπορεί πια να θεωρεί ότι είναι κυρίαρχο κράτος ή δημοκρατία η Μεγάλη Βρετανία. Η Βρετανική λοιπόν κυβέρνηση πρέπει να απορρίψει αυτά τα μέτρα και να προασπίσει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου της. Αλλιώς θα έχει υποκύψει σε πιέσεις από έξω. Πρόεδρος, εντάξει τώρα περνάμε στην έκθεση Φερέιρα, της κυρίας Φερέιρα. Για δύο λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ντόρφμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα, ψήφισα υπέρ τη έκθεσης Φεραίρα, καθώς επίσης και υπέρ του συνολικού πακέτου μέτρων. Θέλω να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία και την εισηγήτρια κυρία Φερέρα να την ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνεργασία στο σύνολο του έτους ε, που συνεργαστήκαμε και να την συγχαρώ για το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Είμαι πεισμένος ότι η έκθεση Φερέρα και έτσι η μακροοικονομική εποπτεία είναι κάτι καινοτόμο, είναι κάτι καινούριο. Στον τομέα του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τίποτα άλλο δεν κάνω, κάναμε από το να δημιουργήσουμε αυτά τα οποία υπήρχαν ήδη. Δεν θεσπίσαμε νέα κριτήρια. Και όταν λέγεται ότι με αυτόν τον τρόπο σε σχέση με την ανάπτυξη που ε, δεν λέει προωθείται. Τότε θα ήθελα αντίστροφα να ρωτήσω γιατί δεν τηρήθηκε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτή που λιγότερο τήρησαν αυτό το σύμφωνο σε σχέση με την ανάπτυξη ήταν σαφές ποιες επιδόσεις είχαν και τώρα πρέπει να δούμε ότι ακριβώς το αντίστροφο θα ισχύει θα σεβόμαστε αυτές τις διατάξεις αυτό το οποίο εμπεριέχει η έκθεση Φερέιρα είναι κάτι το καινοτόμο κάτι το καινούριο θα πρέπει να μας βοηθήσει στο μέλλον έγκαιρα νωρί, έγκαιρα και αυτό είναι το σημαντικό να δούμε τι δεν πάει καλά σε ένα κράτος και να δράσουμε άμεσα αν νωρί έγκαιρα το είχαμε κάνει αυτό στο παρελθόν η Ελλάδα η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία δεν θα είχαν τέτοια προβλήματα. Ήδη προετών θα είχαμε δει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και θα είχαμε κάνει κάτι. Τώρα χαιρόμαστε που αυτό το, αυτός ο μηχανισμός αποτελεσματικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή και να λειτουργεί σωστά η Ένωση και να προασπίσουμε την ευημερία των πολιτών της επίσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το πλήρες ε, πλήσιο της οικονομικής διακυβέρνησης να είναι συμβατά με τις στρατηγικές ε, της Ένωσης για την ανάπτυξη και την ε, απασχόληση με το στόχο να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική σταθερότητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβληθούν κυρώσεις για να τιμωρούνται οι ε, απάτες ε, για να πληρώνονται πρόστιμα και για τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών ε, αγορών. Τα μέτρα που συζητούνται σήμερα έχω το φόβο ότι θα αποδυναμώσουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι η περίπτωση αυτή της έκθεσης Φερέιρα που υποστηρίζει την κοινωνική ισορροπία. Το υπόλοιπο πακέτο όμως δεν πάει καλά γιατί στοχεύει αποκλειστικά στην ε, λιτότητα και δεν προωθεί την ανάπτυξη. Η Ευρώπη θα έχει μέλλον μόνο αν θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, την αυστηρότητα σχετικά με τους λογαριασμούς με τους στόχους της ε, αύξησης και της, απασχόλη... και της ανάπτυξης και της Προέδρο, ευχαριστούμε κύριε Ντάντζελη. Η κυρία Μουσκαρντίνη τώρα Ευχαριστώ πρόεδρε. Η παγκόσμια κρίση ε, έχει υπονομεύσει την ικανότητα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό. Τα μέτρα που υιοθήθηκαν σήμερα με την έγκριση του Six Pack θα βοηθήσουν να προληφθούν οι μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Αλλά πρέπει να βοηθηθούν άμεσα οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό με διάφορους κολέγους, ε, ε, συναδέλφους των πολιτικών ομάδων υποβάλαμε μια πρόταση ψηφίσματος ούτως ώστε η Ευρώπη να προβλέψει ένα μέτρο ε, μια τριετού τους ε, ε, μη φορολόγησης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω από ένα συγκεκριμένο τζίρο και να υπάρχει ε, ε, μια επιδότηση της κοινωνικής ασφάλισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ε, εργαζόμενους. Έτσι θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και θα περιορίσουμε την ανεργία που έφτασε σε απαράδεκτα επίπεδα και καλούμε το Συμβούλιο να προχωρήσει σε τριμερή διάλογο με το Κοινοβούλιο για τις προτάσεις αυτές ευχαριστούμε. Ο τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κανονισμός που ψηφίσαμε για την πρόληψη και διόρθωση των ε, υπερβολικών μακροοικονομικών ισορροπιών μεταξύ των 27 χωρών είναι μια καινοτομία σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Ορίζει κανόνες και ελέγχους και ιδιαίτερα εισάγει την έννοια της συμμετρίας βάσει της οποίας η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογεί όχι μόνο τα ε, λύματα αλλά και τα πλεονάσματα. Στην πράξη, αντίθετα με ό,τι συνήθως πιστεύετε, ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιες χώρες ε, κακές όπως η Ελλάδα ή η Ιταλία, αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα θα τεθούν υπό έλεγχο χώρες όπως και η ε, Γερμανία και η Ολλανδία για το λόγο ότι έχουν πολύ μικρή εσωτερική ζήτηση και εισάγεται μια ομοσπονδιακή προοπτική ε, με βάση την αρχή της ισότητας. Πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά της μελλοντική Ευρώπης και του μέλλοντος των κρατών μελών. Ε, και ε, αυτά είναι οι προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Καρόνα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτίμησα όλο ιδιαίτερο την δουλειά του, της κυρίας Φερέιρα ε, στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Πράγματι, στα πλαίσια αυτού του πακέτου του νομοθετικού που αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, μόνο ε, για αυτή την έκθεση εγώ και η ομάδα μου ψηφίσαμε υπέρ. Διότι μεταξύ άλλων εισάγεται μια ρήτρα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων ε, ξεκινώντας από τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις και υπάρχει και μια ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ε, πράξεις κατανάθεση. Παρόλο που δεν μπορεί να αλλάξει η συνολική ισορροπία του πακέτου των έξι προτάσεων, με την έκθεση αυτή ε, σίγουρα γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός. Ε, διότι εκτός άλλων προβλέπει και ένα σύστημα εποπτείας που λαμβάνει υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια και ε, παρόλο που ε, κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μια οπτική που βασίζεται μόνο στις αρχές της λιτότητας και δεν έχει θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά λέω η έκθεση αυτή είναι μια θετική νότα που πάει αντίθετα προς την τάση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μεσαρός παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. 29 Σεπτεμβρίου 2010 πρότεινε ένα πακέτο μέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον στόχο να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Έξι στοιχεία είχε και έχει και γι' αυτό αποκαλείται six pack και αφορά και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και δύο νέου κανονισμούς που αφορούν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν, πώς πρέπει να εντοπίζονται και να θεραπεύονται. Σε σχέση με αυτές τις προτάσεις ε, υπάρχουν και νέα στοιχεία που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν ε, δείκτες κινδύνου όσον αφορά ανισορροπίες και σε τακτά διαστήματα σύνταξη εκθέσεων αναχώρα. Οι χώρες της Ευρωζώνης που δεν ε, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προτάσεις ε, μπορούν να τεθούν υπό επιτήρηση και να ε, αντιμετωπίσουν και κυρώσεις που ενδεχόμενα μπορούσαν, θα μπορούσαν να επιβληθούν σε αυτές. Όχι μόνο κυρώσεις όμως πρέπει να επιβάλλονται αλλά και κίνητρα πρέπει να δίνονται. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται. Θα πρέπει να επενδύονται σε μακροπρόθεσμα προγράμματα. Η κυρία Χάρκιν παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω στο άρθρο 1 ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής στην Ένωση θα στοχεύει μεταξύ άλλων στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας διότι, και όλες μας, διότι τελικά μόνο έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη μαζί με την οικονομική συνοχή. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου είναι κάτι που, το οποίο επίσης βρίσκω θετικό. Είναι ζωτικό να δημιουργηθεί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Επίσης σημαντικό είναι σε όλες αυτές τις προτάσεις να γίνονται οι συνεννοήσεις δημόσια για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει τι συζητιέται και τι αποφάσεις παίρνονται στο όνομά του. Τέλος συμφωνώ με τον συνάδελφό μου Αυγία ο οποίο είπε ότι η τα πλεονάσματα είναι κοινή ευθύνη όλων μας. Ε, τα ελλείμματα μάλλον. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Α, ο κύριος Σιλβέστρης παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και σε άλλες εκθέσεις, εδώ η ψήφος μας ήταν θετική, διότι η έκθεση αυτή προβλέπει ε, μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών και θεσπίζει κανόνες και εγγυήσεις που λείπουν αυτή τη στιγμή, όπως έδειξε η κρίση ε, και μας δίνει ευθύνε ελέγχου και εποπτείας στην Ευρωζώνη. Μηχανισμοί που είναι ήμι αυτόματη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίκριση που ακούστηκε. Αλλά με κυρώσει ε, που ε, επιβάλλονται ε, για όλες τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που διαπιστώνονται. Αυτό είναι ένα βήμα αποτελεσματικό που θα συμπληρωθεί με επόμενα βήματα που και είναι ίσως συμπτωματικό, αλλά είναι σημαντικό που σήμερα ανέφερε ο πρόεδρος Παρόζο και άλλα μέτρα, ε, όπως ε, φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ε, ούτως ώστε το κόστος της κρίσης να μην το πληρώνουν μόνο οι οικογένειες και η παραγωγή υλικών αγαθών, αλλά και αυτοί που κινούνται στις χρηματοοικονομικές αγορές. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Σιλβέστες. Περνάμε στην έκθεση ΦΕΙΟ. Ο κύριος Ουτζίας παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε για την έκθεση ΦΕΙΟ που αναφέρεται και στην αναθεώρηση του Συμφώνου ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα χρόνο αργότερα μετά την αρχή υποβολή της πρότασης. Προβλέπεται ένας έλεγχος ε, στα κράτη-μέλη που έχουν ε, σχέση 60% ή παραπάνω, ε, μία μείωση χρέους δηλαδή ΑΕΠ πάνω από 60%, μία μείωση 50%. Είναι ο ρυθμός που έχει σημασία εδώ για την μείωση αυτή. Η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη της μία ολόκληρη σειρά από χαρακτηριστικά πριν κάνει τις συστάσεις της στο κάθε κράτος μέλος. Εισάγεται η βασική αρχή ότι μειώνοντας το χρέος ε, χρειάζεται να πληρώνονται λιγότεροι τόκοι και έτσι δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα κονδύλια για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη που είναι ο πραγματικός στόχος επί του οποίου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας κατά τους προσεχείς μήνες. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέρφυ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένας από τους στόχους μας εδώ είναι να δρούμε ως δημοκρατική πρόσωψη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κυριαρχείται από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Αυτή η πρόσωψη όμως ακόμη και αυτή αρχίζει να καταστρέφεται σήμερα γιατί δεχτήκαμε την εξάμετρο που τελικά θα δώσει περισσότερες εξουσίες στην Κομισιόν για να δράσει ως χωροφύλακας της λιτότητας. Έτσι ελήφθησαν επίσης μέτρα ώστε μία απλή πλειοψηφία στο Συμβούλιο να μην μπορεί να περάσει την καταδίκη τέτοιων μέτρων. Περιορισμένη δημοκρατία λοιπόν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία περιορίζεται ακόμη περισσότερο με αυτή την προσπάθεια να επιβληθεί η λιτότητα. Τι φοβάται η Κομισιόν, φοβάται την εργατική τάξη και το εργατικό κίνημα της ε, εξεγέρσης στην Ελλάδα, στην Ισπανία και αυτά τα κινήματα και ιδίως φοβάται μήπως συνδεθούν και συνδυαστούν. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρκιν παρακαλώ. Συμφωνώ με το σημείο 4α που λέει ότι ο κανονισμός αυτός δεν αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση άμεσα, αλλά περισσότερο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη και κοινωνική προσέγγιση. Πολλέ φορέ είπα σήμερα ότι δεν προτείνουμε λύσει για την τρέχουσα κρίση, αλλά μια δυνατότητα που προβλέπει αυτή η έκθεση θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση με την επίτευξη μια ολοκληρωμένη και δυναμική εσωτερική αγορά. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει σημαντική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα αυτό έχει μεγάλε επιπτώσει για τη χώρα μου, την Ιρλανδία. Χαίρομαι που αναφέρεται ότι οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι των χωρών που προσπαθούν να ε, επιτύχουν αριθμό ανάπτυξης θα ληφθούν υπόψη. Και γίνονται, όταν θα γίνονται προτάσεις ε, στα κράτη-μέλη για διορθωτικά μέτρα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό είναι ένας τρόπος επίτευξης εσωτερικής ε, σύνοχης και επίσης υπάρχουν συστάσεις για σεβασμό του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για την υποστηρίξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Θα περάσουμε στην έκθεση Ford τώρα. Θα λάβει τον λόγο ο κύριο Μπαλταζάρε, παρακαλώ. Πρόεδρε, η περιοδική διαθεσιμότητα ε, αξιόπιστων ε, δεδομένων ε, των δημοσιομικών των κρατών μελών είναι ένας παράγοντας κλειδί για να λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα σε περίοδους κρίσης. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει η Κομισιόν να μπορεί να εποπτεύει τη συμβατότητα με τους κανόνες του προβολισμού των κρατών μελών. Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι βάσει της συνθήκης ε, η θέσπιση ενός μεσοπρόσωσμου δημοσιονομικού πλαισίου δίνει τη δυνατότητα ε, στις διάφορες κυβερνήσεις να τροποποιούν και να προσαρμόζουν τις προηγούμενες επιλογές. Είναι απαραίτητο λοιπόν η οδηγία αυτή να εφαρμοστεί πιστά και η Κομισιόν να εποπτεύει ε, συστηματικά την εφαρμογή της, ούτως ώστε να αποφύγουμε να έχει απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο της οδηγίας δηλαδή μια ομοιόμορφη, ε, ένα ομοιόμορφο σεβασμό ε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως το απαιτεί η συνθήκη. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ουτζίας παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω από ένα χρόνο πριν όταν ε, άρχισαν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και μετά και των άλλων χωρών, έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ευρωπαϊκό κανάλι. Και ένα από τα θέματα που έθιξα ήταν ακριβώς το θέμα των στατιστικών στοιχείων που επέτρεψαν σε κάποιες χώρες να μαγειρέψουν τους λογαριασμούς και έτσι με την έκθεση Ford που υπερψηφίσαμε σήμερα εισάγονται αντίθετα κριτήρια διαφάνειας και ανεξαρτησίας των εθνικών στατιστικών αρχών με κυρώσεις που προβλέπονται για αυτούς που ε, ε, μαγειρεύουν, παραποιούν τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, διότι στοχεύει στην έλλειψη διαφάνειας των στατιστικών στοιχείων και τα καθιστά ομοιόμορφα. Και αυτό θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και στις ε, εθνικές κυβερνήσεις να προχωρούν ε, με κοινό βήμα, γνωρίζοντας ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε κυρία Χάκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστήριξα την έκθεση αυτή και δέχομαι ιδιαίτερα αυτό που λέει ότι μια ολοκληρωμένη λύση για την κρίση των χρεών στην Ευρωζώνη πρέπει να συνδυαστεί. Σήμερα θεσπίσαμε ένα τμήμα της λύσης των μέτρων η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι κάτι το ουσιώδες και ο Επίτροπος Ρεν πρότεινε και περισσότερη αλληλεγγύη μέσω των ευρωμολόγων. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν και άλλες λεπτομέρειες να συνδυαστούν, να συνοδευτούν όλα αυτά τα μέτρα και με περισσότερα. Το, ο πολιετής δημοσιονομικός σχεδιασμός δεν εμποδίζει καμία εκλεγμένη κυβέρνηση από το να μετατρέψει η προηγούμενη πολιτική της. Τέλος, οι εκθέσεις αυτές αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που αφορά 17 χώρες μέλη. Αν μία έχει νομισματικό πρόβλημα, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε, πρέπει να το λύσουμε με τρόπο δίκαιο και επαρκή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κυρία Χάκιν. Κυρία Χάρκιν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εσείς και ο κύριος Ουτζίας σήμερα πραγματικά είσαστε άξιοι του μισθού σας. Δουλέψατε πολύ. Και περνάμε αμέσως στις τελευταίες επεξηγήσεις, τελευταία επεξήγηση ψήφου για την έκθεση για τις προτάσεις ψηφίσματος για το γενετήσιο προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου. Έχει τον λόγο κυρία Ματσόνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό ε, αναφέρεται στη δήλωση της κυρίας Άστον ε, κατά την ε, Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας. Με τη δήλωσή της η Κάθριν Άστον επανέλαβε την δέσμευση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων υπέρ όλων των δράσεων που καταπολεμούν τη βία απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού του και της ταυτότητας φύλου. Ε, είμαι ικανοποιημένη που με αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κάνει το ίδιο. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω ότι η υπερψήφιση του ψηφίσματος αυτού εκ μέρους μου σκιάζεται από μία μόνο αμφιβολία. Δηλαδή στην παράγραφο 11 θα ήθελα να ε, ε, ε τροποποιηθεί ε, διότι κάποιες ε, πολιτικές ομάδες εισάγουν λανθασμένες έννοιες. Ε, αναγνώριση δικαιωμάτων που φορούν την οικογένεια. Αυτό είναι λάθος, γιατί αυτό δεν είναι αρμοδιότητα αυτού του θεσμικού οργάνου. Αυτή τη στιγμή που θέλουμε, από τη στιγμή που θέλουμε να καταπολύσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας, δεν μπορούμε να μιλάμε τέτοια. Κυρία Τσέσκοβα, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπεψήφισα, ψήφισα υπέρα της της πρότασης ψηφίσματος για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν οι γενετήσιες επιλογές και η ταυτότητα φύλου εξακολουθούν να είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτοί που ανήκουν σε αυτές τις μειονότητες είναι πολλές φορές ε, θύματα αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης και κακομεταχείρισης και πρέπει να μεριμνήσουμε και να δούμε ότι αυτό δεν θα είναι μόνο θέμα ποινικών διαδικασιών και ε, εγκληματικών διώξεων αλλά και πολλές φορές θέμα ε, της ε, ίδιας της δίωξης και της θανατικής ποινής και πάσης φύσεως στρεβλών πρακτικών. Θα έπρεπε όλα τα άτομα να έχουν τα ίδια δικαιώματα χωρίς αρνητική μεταχείριση. Γι' αυτό Καλοχαιρετίζω το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που είναι το πρώτο αυτού του είδους και που αφιερώνεται στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και αποδεικνύει την οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα έπρεπε να υποστηρίξουμε τη διεξαγωγή ενός διαλόγου σε αυτόν τον τομέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε σε όλες τις δραστηριότητες να έχει μια ενιαία κοινή στάση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Και μια στιγμή, ποιος θα πάρει το χρυσό, κύριο Σιλβέστρης παρακαλώ. Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ των ε, συναδέλφων που καταψήφισαν αυτή την πρόταση. Όχι γιατί δεν ε, συμφωνώ φυσικά την ε, ε, καταδίκη της ομοφοβίας ή την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πρώτη που θα πρέπει να σεβαστεί το δικό της χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων, αλλά γιατί αντίθετα θεωρώ ότι όταν είπε και η συνάδελφος Ματζόνη, όταν ε, λέγονται αυτά που λέγονται στην ε, παράγραφο 11, είναι μια υπόγεια προσπάθεια να αρνηθούμε όλα αυτά που που υποστηρίζουμε. Διότι κάθε φορά που ε, αναφερόμαστε ε, με οποιοδήποτε τρόπο στο θέμα της αναγνώρισης του ε, φίλου, της ταυτότητας φίλου, υπάρχουν κάποιοι που για πολιτικούς σκοπούς ή γιατί θέλουν να περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια νομοθεσία που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν όπως νομίζουν και άλλα φύλλα εκτός από το αρσενικό και το θηλυκό, προσπαθούν να περάσουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ε, δεν ε, Δεν πρόκειται για μια Ευρώπη που θέλει να αλλάξει τους νόμους της φύσης που μας έκανε άντρες και γυναίκες. Απλώς Πρόκειται για μια προσπάθεια εξασφάλισης των πολιτικών δικαιωμάτων του ε, καθενός και όχι ε, να περνάνε μέσα από τα θέματα του φίλου επιχειρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Γι' αυτό με μεγάλη μου δυσαρέσκεια καταψήφισα αυτή την πρόταση. Ολοκληρώθηκαν οι επεξήγησεις ψήφου και θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα με τις εργασίες στην Ολομέλεια. Γεια σας.